χρησιμοποιήσουμε σωστά και έξυπνα για να αποκομίσουμε τη σωστή προστιθέμενη αξία και να βοηθήσουμε τους πολίτες, τα 160 εκατομμύρια πολιτών που ζουν κατά μήκο του Δούναβη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Κλείνει η συζήτηση το θέμα αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει την 5η το μεσημέρι στις 12. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η δήλωση της Επιτροπής για τα βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος. Ο κύριος Ντάλι. And whenever you are ready, Commissioner, you have the floor. Όποτε είστε έτοιμος, κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. President, honorable members. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, η επιστημονική πρόοδος στις τελευταίες δεκαετίες συνέβαλε σε αυξημένη χρήση των ε, ε, κυτάρων, κιτάρων κυτάρων από φαλικό αίμα και των σχετικών φαρμάκων. Αυτό είχε θετικά αποτελέσματα για ασθενείς με διαταραχές αιματολογικές όπως η λευχαιμία. Αυξημένη χρήση των ε, βλαστικών αυτών κυτάρων θα μπορούσε να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε και άλλες ασθένειες γενετικού χαρακτήρα. Ε, και τα ενήλικα βλαστικά κύτταρα έχουν σημαντική ε, δυνατότητα ε, αξιοποίησης. Όμως χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για τις δύο αυτές κατηγορίες κυτάρων. Η μεταμόσχευση πλαστικών κυτάρων εμπεριέχει τον κινδυνό μετάδοσης κάποιων ασθενειών. Γι' αυτό πρέπει να θεσπιστεί ένα νομικό πλαίσιο για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της χρήσης των ε, ανθρώπινων βλαστικών κιτάρων. Για τους σκοπούς αυτούς πρέπει όμως να ξεκαθαρίσω κάτι. Τα κράτη-μέλη από μόνα τους αποφασίζουν για το πώς και εάν θα χρησιμοποιήσουν τα βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για την εναρμόνιση της χρήσης των βλαστικών κυτάρων. Ε, ε, σχετικές οδηγίες ε, αναφέρουν ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παρεύει στην χρήση ή μη χρήση ο, κατά οποιονδήποτε τρόπο των βλαστικών κυτάρων ομφαλικού αίματος. Αν όμως τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τα βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος, αυτό θα πρέπει να πληρεί τις απαιτήσει ε, ποιότητας και ασφάλειας της οδηγίας, δηλαδή προστασία της δημόσιας υγείας και ε, σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουν ε, ακριβή ενημέρωση οι πολίτες όσον αφορά τα πλεονεκτήματα και τους κινδύνους της χρήσης των βλαστικών κοιτάλων. Η παροχή ε, αυτή της ενημέρωσης και πάλι είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να πάρουν τα σχετικά μέτρα και κάποια το έχουν ήδη κάνει. Τέλος θα πρέπει να σε βεβαιώσω ότι η Κομισιόν τακτικά παρακολουθεί ε, την ε, μεταφορά της σχετικής οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο των κρατών μελών και ε, αυτό σε σχέση με την οδηγία που ε, συζητήθηκε στον, στο Κοινοβούλιο πέρυσι τον Ιανουάριο. Ευχαριστώ οι πολιτικές ομάδες και πρώτος ο μιλητής ο κύριος Λίζα εκ του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ε, χαίρομαι που βρήκατε το χρόνο έστω και αργά να έρθετε εδώ και να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έρευνα στον τομέα των βλαστικών κυτάρων παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες ε, για ασθενείς, τους οποίους δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε μέχρι τώρα. Μιλάμε και για βασική έρευνα, αλλά μιλάμε για ασθένειες, ε, ε, ε, για πάνω από 70 ασθένειες, στις οποίες μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς με τα βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος. Τα βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος γίνονται, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή κυρίως από αλλογενή δημοσιεύματα και μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε τέτοια κύτταρα στη Λευχαιμία, παραδείγματο χάρη, ε, για παιδιά που δεν, μπορούν, ε, δεν μπορεί ο οργανισμό του να σχηματίσει αυτά τα κύτταρα. Υπάρχουν πολλέ μορφέ θεραπεία από τι οποίε μπορούμε να υποφεληθούμε ευρύτατα σήμερα. Και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξουν τα κατάλληλα πολιτικά μέτρα, ούτω ώστε να υποστηρίξουμε τι δημόσιε τράπεζε για βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Αλλά θα πρέπει παράλληλα να βοηθήσουμε και ε, να μην απαγορεύσουμε την αυτόλογη ε, μεταμόσχευση και τα αντίστοιχα μέτρα. Θα πρέπει δηλαδή η πολιτική να είναι ενημερωμένη για τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Θέλουμε σαφή πρότυπα ασφάλειας και ε, να γίνεται σωστή χρήση των βλαστικών κιτάρων, να τηρούνται τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας, ούτως ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μέχρι τέλους αυτά τα κύτταρα τα οποία λαμβάνονται. Και θα πρέπει να φροντίσουμε να μπορούν να αποφασίζουν οι γονείς για το ότι δεν θέλουν να πετάξουν τα βλαστικά κύτταρα του ομφαλικού αίματος γιατί ίσως είναι κάτι το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε για το δικό τους παιδί είτε για άλλα παιδιά στο μέλλον αν αποθηκεύσουν το ομφαλοβλακουντιακό αίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λίζε. Η κυρία Ρή, εκ μέρους των, των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου και κυρίως τον κύριο Λίζε και τον Λουίς Πέτερλε που είχαν αυτή την ευτυχή πρωτοβουλία να μιλήσουμε για τα βλαστοκύτταρα του ομφαλικού αίματος. Πρόκειται για μια τρομερή πρόοδο εδώ και 20 χρόνια με την ε, μεταμόσχευση που επιτυγχάνεται και έτσι μπορούν να θεραπευθούν κυρίως ε, γύρω στα 80 νοσήματα όπως λεμφώματα, ανεμίες, αυτόνες ονομήματα, σπάνιες ασθένειες, λευχαιμία κτλ. κτλ. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω ότι μόνο 1% αυτού του τόσο πλούσιου αίματος από τον Πλακούντα ε, κρατείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1 εκατομμύριο με 15 εκατομμύρια γεννήσεις ε, ετησίων ε, γι' αυτό θα πρέπει να ζητήσουμε την Επιτροπή να κάνει σε συνεργασία βεβαίως και το υπενθύμησε ο Επίτροπος με τα 27 κρατικά μέλη μία εκστρατεία προς τους μελλοντικούς γονείς ώστε η δωρεά ε, βλαστοκυτάρων από τον ομφάλιο λόρο να γίνει ε, κάτι το προφανές. Πιστεύω λοιπόν ότι εκτός από την μεταφορά της οδηγίας του 2004 για την ασφάλεια ιστών και κιτάρων, πράγμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, πιστεύουμε ότι είναι έχει σημασία να ενθαρρύνει πάρα πολύ τα κράτη-μέλη Ευρωπαϊκή Ένωση να απλωστεύσουν το θέμα της διαπίστευσης των μευτηρίων που είναι σε δυνα... έχουν τη δυνατότητα να ε, φυλάξουν σε ασφαλείς συνθήκες τα βλαστικά ε, κύτταρα καθώς και να διασφαλίσουν την χρησιμοσύπησή τους. Εδώ, όπως είπε και ο κύριος Επίτροπος, δεν θα πρέπει να υπάρχει γενικότερη αποσιώπηση του τρόπου με τον οποίο αποθηκεύεται τα, ε, αποθηκεύονται τα βλαστοκύτταρα αλλά να γίνουν τα βλαστοκύτταρα από τον ε, ομφάλιο λόρο δωρεά ζωής. Ευχαριστώ. Εκ μέρου των Πρασίνων... Η κυρία Άουκεν, εκ μέρου των Πρασίνων. Και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να δημιουργηθούν τέτοιες τράπεζες για τα βλαστικά κύτταρα ομφαλικού αίματος δεν θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία όπως ε, στις μεταμοσχεύσεις. Θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία στην οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αίμα κατά τον ε, ε, σωστό τρόπο, έχοντας λάβει τα απαραίτητα μέτρα και πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, όπως αυτά που ανέφερε ο κύριος Λίζε. Υπάρχουν πολλέ δυνατότητε και ίσω ακόμη να υπάρχουν και άλλε δυνατότητε τι οποίε δεν γνωρίζουμε ακόμη και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιε τράπεζε. Θα πρέπει να είναι ανοιχτή η πρόσβαση σε αυτέ τι τράπεζε και να μπορούν να τι χρησιμοποιήσουν όλοι. Και ε, επίσης ε, είναι σημαντικό ε, να αποφύγουμε τις πιθανές παγίδες. Παραδείγματος χάρη, πολλές φορές προσπαθούν να πείσουν τους γονείς να πληρώσουν ε, ε, περισσότερα χρήματα για την ασφάλεια των παιδιών τους ούτως ώστε ε, για να διατηρηθούν τα κύτταρα αυτά θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερα χρήματα οι γονείς. Πρέπει σε όλα τα επίπεδα να λάβουμε λοιπόν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας να είναι ανοιχτή η πρόσβαση και να έχουμε σωστά ε, πρότυπα. Σε αυτά θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι οι γονείς μπορεί και να εξαπατώνται ή μπορεί και να φοβούνται ότι δεν θα επενδύσουν επαρκώς στην ασφάλεια του παιδιού τους στο μέλλον εάν δεν υποκύψουν ε, σε αυτές τις προσφορές. Ε, γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε τα σωστά μέτρα σε όλους τους τομείς. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Άουκεν. Η κυρία Μαρίσα Ματίας εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να πω ότι πιστεύω ότι το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να συνεχίσουμε να ζούμε ε, χωρίς ε, τις ψευδείς υποσχέσεις τις οποίες είχαμε μέχρι τώρα στην Ευρώπη, κυρίως όσον αφορά την συλλογή των βλαστικών κιτάρων του εμφαλικού αίματος. Πολλές φορές υπάρχουν βάσεις δεδομένων οι οποίες οδηγούν σε απάτες. Ε, είπε η συνάδελφος ότι οι δυνατότητες τέτοιου είδους δωρεών φτάνουν μόνο στο 1%. Ξέρουμε ότι παρόλα αυτά θεραπεύουν πάρα πολύ σπάνιες ασθένειες και σοβαρές ε, τα βλαστικά κύτταρα όπως το Αλσχάιμερ και οι ε, διάφορες μορφές καρκίνη. Θα πρέπει να πούμε σε όλους, στις μητέρες και στους πατέρες ότι μπορούν να κρατήσουν τα βλαστοκύτταρα των παιδιών τους από τη γέννησή τους και να μπορέσουν αν είναι ε, στο μέλλον αναγκαίο να θεραπεύσουν τα παιδιά τους από κάποια ασθένεια. Πολλοί το είπαν αυτό. Αυτό ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ λανθασμένη υπόσχεση. Στην ποτοργαλία αυτή η ψευδής υπόσχεση για την ε, ε, διαφύλαξη των κιτάρων σε ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης κοστίζει 3 και 4 μισθούς στο μέσο Πορτογάλο. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότητα μεταξύ όλων, να υπάρχουν δημόσιες τράπεζες φύλαξης και να υπάρχουν ε, χρησιμοποίηση για όλους και για όλες τις ασθένειες και όχι για μόνο ολίγους. Πιστεύω λοιπόν ότι η αμερόληπτη ενημέρωση ε, συνεργασία και αλληλεγγύη είναι η καλύτερη λύση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να επιβάλλουμε τίποτε. Μπορούμε όμως εξ ονόματος ισότητας να δημιουργήσουμε κίνητρα ώστε να γίνει επωφελής ε, για όλους αυτή η διαδικασία. Κύριος Πέτρα. Κύριε Επίτροπε, χαιρετίζω την ε, πρόθεσή σας υποστηρίξετε αυτό το οποίο κάνουμε εδώ. Νομίζω ότι με αυτή την πράξη θα προσεγγίσουμε περισσότερο και τους πολίτες. Όπως είπαν και οι συντάκτες. Νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό το θέμα με όλα αυτά τα οποία κάνουμε και για τα οχήματα. Νομίζω ότι το θέμα αυτό ενδιαφέρει και απασχολεί όχι μόνο τους μελλοντικούς γονείς αλλά όλους όσους ασχολούνται με τις εφαρμογές ε, των βλαστικών κιτάρων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει κάποια μέτρα. Βλέπουμε ότι προς το παρόν αυτά τα βλαστοκύτταρα τα οποία χάνονται θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή συνεργασίας και θεραπείας. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους γονείς κάνοντας τη σωστή ενημέρωση και να πείσουμε τους πολίτες ότι κάνουμε ό,τι κάνουμε προς την ε, σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Περνούμε τώρα στις παρεμβάσεις διαρκείας ενό λεπτού και πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο στον κύριο Καντσιέν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Πιστεύω ότι το θέμα αυτό, έστω και αν είναι αργά το βράδυ, είναι ένα σημαντικό θέμα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη γιατί πιστεύω ότι η θεραπευτική χρήση των βλαστοκυτάρων ομφαλικού αίματος είναι κάτι που θα πρέπει να υποστηριχθεί. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι ε, πρωτοβουλίες και οι ενημερωτικές εκστρατείες ώστε να γίνεται δωρεά ε, του, ε, των βλαστικών κυτάρων και οι, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να δοθούν σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στο ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Είπατε ότι δεν είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα αυτή. Αλλά η μεταφορά της οδηγίας 23 του 2004 ε, δεν καθορίζει κανόνες ποιότητας και ασφάλειας για την ε, ε, συλλογή, τη φύλαξη, τη μεταφορά των κιτάρων. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια συνεκτική πολιτική των συντονισμένη εφαρμογή των εθνικών πολιτικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν τα ίδια δικαιώματα και να υπόκειται στους ίδιους τους νόμους. Επίσης δεν θα πρέπει να συντονιστούν οι εθνικές και ευρωπαϊκές ε, τράπεζες ε, φύλαξης ώστε να ε, διαχειρίζονται με αποτελεσματικό τρόπο όλους τους πολίτες που έχουν αυτές τις ανάγκες. Να καταργήσουμε την ομερτά και να εξασφαλίσουμε τα ίδια δικαιώματα για όλους τους πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάλι έχει τον λόγο. Κέλλη, με συγχωρείτε. Κάνει. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κέλλη. Ε, το θέμα αυτό είναι πολύ αμφιλεγόμενο στην Ιρλανδία. Αυτή τη φορά στις ε, εκλογές Φυσικά η οικονομία κατέχει το κεντρικό ρόλο, αλλά και η ιατρική επιστήμη συζητιέται ε, πάρα πολύ. Και η ποιότητα της ιατρικής έρευνας που έχουμε στα διάφορα ε, Ινστιτούτα ε, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και η ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι γιατροί. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της πρόοδου που έχει πραγματοποιηθεί και έχει υποθεί ότι η πρόοδος αυτή μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε κάποιες συγκεκριμένες ασθένειες και θα πρέπει να ενθαρρυνθεί αυτό το είδος ε, ε, της ε, έρευνας και φυσικά τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μέσα στα πλαίσια της, των περιορισμών της δεοντολογίας. Όπως είπε η Κομισιόν, είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών βεβαίως το κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι αυτοί και το θέμα θα πρέπει να παρακολουθεί εν χρόνο. Ευχαριστώ, κυρία Σίνκλερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, πολλοί συνάδελφοι ήδη σχολίασαν, αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητηθεί όχι μόνο εδώ στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όσο το δυνατόν ευρύτερα. Είναι ένα θέμα που και εγώ ίδια ε, δεν είμαι βέβαια πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ανάμεσα στην καθολική μου προέλευση και στη σύγχρονη επιστημονική κοινότητα πρέπει να, να αποφασίσουμε ποιο δρόμο θα ακολουθήσουμε. Έχετε δίκιο κύριε Επίτροπε σε αυτό που είπατε. Είναι κάτι που πρέπει να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη οι πολιτιστικές και θρησκευτικέ διαφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνουν σεβαστές και δεν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πάρουμε εμείς από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σίγκλερ. κύριος Μικολάσιτς. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω δύο λόγια για τα πλαστοκυδάρα αμφαλικού αίματος. Η συλλογή ε, ομφαλικού αίματος κατά το τοκετό που μέχρι τώρα πεταγόταν στα σκουπίδια μπορεί να είναι μια σημαντική πηγή μη διαφοροποιημένων βλαστοκυτάρων που μπορούν να τροποποιηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στο μέλλον και να χρησιμοποιηθούν για την μετώπιση καρκίνου και άλλων ασθενειών, τουλάχιστον 70 διαφορετικών ασθενειών και από ό,τι ξέρω λιγότερο από το 1% ε, του ομφαλικού αίματος συλλέγεται στην Ευρώπη. Και είπε η Κομισιόν ότι είναι θέμα των κρατών μελών να ρυθμίσουν αυτή την υπόθεση, αλλά η Κομισιόν θα μπορούσε να βοηθήσει με παροχή πληροφοριών προς τους γονείς σχετικά με τα πλεονεκτήματα των βλαστοκυτάρων και την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί σε αυτόν τον ερευνητικό τομέα και στον τομέα αυτό της επιστήμης. Ε, το λέω αυτό ε, ως ε, τέος εισηγητής για την πρόοδο των θεραπευτικών μεθόδων. Ο τελευταίος ομιλητής για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την συμβολή της στο θέμα αυτό. Όμως λόγω των ανησυχιών που εκφράστηκαν, ίσως μια λύση θα μπορούσε να είναι τα εθνικά μητρώα των τραπεζών αίματος θα να χρησιμοποιηθούν σαν μητρώα και για την φύλαξη ε, βλαστικών κυτάρων ομφαλικού αίματος για μελλοντική χρήση. Αυτό θα μπορούσε να λύσει κάποιες από τις δυσκολίες που ανέφεραν οι συνάδελφοι όσον αφορά το κόστος της αποθήκευσης. Εφόσον έχουμε ένα σύστημα ήδη που λειτουργεί για τις εθνικές τράπεζες ε, ε, αίματος, αυτό το σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει για τον έλεγχο της ποιότητας και των βλαστοκυτάρων. Αυτό θα μπορούσε να λύσει κάποιες δυσκολίες. Πολλοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι υπάρχουν πολύ σημαντικές προοπτικές για την χρήση των βλαστοκυτάρων στο μέλλον για αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών. Θα πρέπει να προσέξουμε όμως να μην δημιουργούμε και ψευδείς ε, ελπίδες, γιατί πολλές φορές και σε άλλους τομείς έχουν δοθεί ψεύτικες ελπίδες στον κόσμο. Πρέπει να ε, ε, έχουμε λοιπόν ε, επιστημονικές αρχές και να έχουμε επιστημονικά αποτελέσματα για να μπορούμε στη συνέχεια να ισχυριστούμε ότι έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Ντάλη για να συνοψίσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Αναμφίβολα υπάρχει γενικότερη λόγηση της πρόοδρου η οποία έχουμε για την ε, χρησιμοποίηση των βλαστοκυτάρων για θεραπευτικούς λόγους. Συμφωνούμε ότι όντως θα πρέπει να ενθαρρυνθεί αυτή η πρακτική. Τα θέματα που ανέφεραν οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτές όντως είναι θέματα ενημέρωσης και αποθήκευσης. Όσον αφορά την ενημέρωση, είναι σημαντικό και συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να παρέχεται η σωστή ενημέρωση στους γονείς και σε όλο τον κόσμο γενικότερα για την ε, χρησιμοποίηση των βλαστοκυτάρων, κυρίως των βλαστοκυτάρων του ομφαλίου λόγου. Αυτό είναι ένα θέμα αρμοδιότητας των κρατών μελών. Πολλές φορές όμως ξέρουμε ότι κάθε ε, κράτος διαφέρει ως αναφορά την χρησιμοποίηση, τα μειονεκτήματα και τους περιορισμούς των βλαστοκυτάρων. Πολλά κράτη-μέλη ήδη έχουν συστήσει εκστρατείε ενημέρωση και άλλε δραστηριότητε. Η Επιτροπή ενθαρρύνει ε, τα κράτη-μέλη να λαμβάνουν τέτοιου του δράσει. όσον αφορά την αποθήκευση. Γνωρίζουμε ότι οι ιδιωτικές εταιρείες ήδη προσφέρουν στου γονεί ε, την υπηρεσία αυτή της φύλαξης και της αποθήκευσης των βλαστοκυτάρων. Παρ' όλα αυτά, πολλά κράτη-μέλη έχουν δημόσιες τράπεζες φύλαξης βάσει ε, δωρεών, αλτρουιστικών και δωρεάν. Ξέρουμε ότι η σχετική οδηγία περιστών και κιτάρων θέλει να θεσπίσει τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν σε ιδιωτικό και ε, δημοσιοπίπεδο βάση βάσει της ανωνυμίας, της ε, αλληλεγγύης μεταξύ δότη και αποδεχόμενη. Ξέρουμε ότι η θα πρέπει να δημιουργηθούν δημόσιες τράπεζες ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση δωρεάν όλοι οι ασθενείς σε τέτοιου είδους βλαστοκύτταρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Η συζήτηση αγαπητοί συνάδελφοι για τα βλαστοκύτταρα εμφαλικού αίματος ολοκληρώθηκε. Έχουμε ακόμη ένα θέμα στην ημερήσια διάτοξη. Τις παρεμβάσεις διαρκείας ενός λεπτού σύμφωνα με το άρθρο 150 του κανονισμού